Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν τα έχει κάτσει και ο συνάδελφος με το κινητό του. Λοιπόν, συμφωνήσαμε την τελευταία φορά ότι δεν θα τυπώνουμε τα έγγραφα παρά μόνο για ειδικού προσκεκλημένους και με τον τρόπο αυτό εξοικονομήσαμε χρήματα, χρόνο, χαρτί. Εσύ δεν το έχει ζητήσει αυτό. Λυπάμαι που το ζήτησε εσύ, αλλά δεν πειράζει, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας την ημερήσια διάταξη και αν δεν <laughs> υπάρχουν αντιρρήσεις, ο κύριος Πίτερ Φαντάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, έχω κάτι να πω που αφορά την ημερήσια διάταξη. Αύριο στις 12.30 με μία παρατέταρτο το Ερευνητικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια θα εκδώσει τα απορίσματά τους όσον αφορά την κατάρριψη, την πτώση του στην Ουκρανία. Είχαμε μια ακρόαση με όλους τους εμπειρογνώμονες πέρσι και στις συνεδρίες των συντονιστών αργότερα ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο ούτω ώστε ο πρόεδρος του ερευνητικού αυτού συμβουλίου να έρθει εδώ και να μας εξηγήσει ποια είναι τα πορίσματα της έκθεσης Ίσως μπορούμε να το οργανώσουμε για τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Ήθελα να το επισημάνω απλώ, ούτω ώστε να βρούμε κάποιο χρόνο να το κουβεντιάσουμε λίγο. Okay, das wäre also nicht für Πολύ ωραία. Αυτά βέβαια ε, δεν αφορούν ε, την ε, σημερινή συνεδρία, αλλά τι συνεδρία του Νοεμβρίου. Θα το κουβεντιάσουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών και θα ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών 14-15 Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τα πρακτικά εγκρίνονται. Πάμε τώρα στο τρίτο σημείο της σημερινής διάταξης. Είναι η παροχή υπηρεσιών στα λιμάνια. Ο κύριος Φλέκενστάν, εισηγητής, και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, 212 ε, τροπολογίες, εκτός 90 ε, δικές μου, άρα οι υπόλοιπε είναι 610 που έχουν ε, κατατεθεί από τους αδέλφους. Αν αυτό δεν είναι επιμέλεια και εργατικότητα, τότε τι είναι. Το σχέδιο των, συμβασμών έχει σταλεί στους και τους για πρώτη φορά, εξετάσαμε τα άρθρα 1 έως 9 αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε σε λογικό συμπέρασμα σε όλες τις περιπτώσεις, απλά εξετάσαμε όλες τις ε, τροπολογίες. Η επόμενη συνάντηση είναι την 5η και η τρίτη συνάντηση έχει προβλεφθεί για τις 27 Οκτωβρίου. Όσον αφορά τώρα στο περιεχόμενο, πρόσβαση στην αγορά και οργάνωση των υπηρεσιών, είναι καθοριστική σημασίας όχι μόνο το ότι αλλάξαμε τις επικεφαλίδες, αλλά θα αλλάξουμε και το περιεχόμενο. Δηλαδή δεν πρόκειται πλέον για την πρόσβαση στην αγορά, αλλά πρόκειται για την οργάνωση των υπηρεσιών των λιμένων. Με τις αλλαγές στο κεφάλαιο 2 θεωρώ ότι πλέον υπάρχει δυναμισμός, μια θετική εξέλιξη και αυτό θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Όλες ε, οι πολιτικές ομάδες στηρίζουν αυτή την προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχει πολυμορφία στην οργάνωση των υπηρεσιών και όχι να ξανακάσουμε τους πάντες να κατέβουν στην αγορά. Όσον αφορά τώρα τη διαφάνεια, αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της έκθεσης και σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις. Αυτά τα δύο θα πρέπει να τα εξετάζει κανείς από κοινού. Η διαφάνεια ε, της ε, αποζημίωσης για παροχή υπηρεσιών στους λιμένες θα πρέπει προφανώς και αυτή να είναι ε, διαφανής κυρίως όταν πρόκειται όταν εμπλέκονται δημόσιοι φορείς αυτό είναι δικαίωμα και απέτηση των φορολογουμένων η διαφάνεια της αποζημίωσης για θέματα υποδομής ε, καταλήξαμε στο ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό της ε, αποζημίωσης ε, θα πρέπει να είναι διαφανή. Στα λιμάνια όμως θα πρέπει επίσης να υπάρχει περιθώριο για ατομικές διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τώρα την ατομική διαφάνεια, πρέπει να αναφέρουμε εδώ τις κρατικές ενισχύσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτές δεν είναι άμεσα με αυτό το κανονισμό, αλλά έμεσα. Και το σχέδιο για την αναθεώρηση του κανονισμού εγκρίθηκε για το τέλος του 2015. Ακούσαμε όμως ότι μέχρι τότε δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Ε, εκεί λοιπόν πρέπει να περιλαμβάνονται τα λιμάνια. Και κατά τη δική μου άποψη ε, στην επόμενη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών θα πρέπει να σκεφτούμε πού είναι οι κόκκινες γραμμές για μας. Και όχι μόνο από πλευράς περιεχομένου, αλλά και από πλευράς διαδικασίας. Δηλαδή, αν ε, όλα αυτά σημαίνουν το διατυπώνω περισσότερο ως ερώτημα. Είναι δυνατόν να υπάρξει μία σαφής δήλωση η οποία θα μας βρίσκει σύμφωνους. Μπορούμε να ψηφίσουμε εδώ, στην Επιτροπή. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας όσον αφορά τη διαδικασία. Και βεβαίως και πρέπει να συζητήσουμε για το περιεχόμενο, αλλά όλοι μαζί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο ένα μικρό κύκλο ατόμων. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση και τις ε, κοινωνικές προδιαγραφές, δεν διαφωνούμε ότι και αυτό θα πρέπει σε επίπεδο αρχής να αναφέρεται, όμως αυτή τη στιγμή διαφωνούμε ακόμα για το πώς θα τα διατυπώσουμε όλα αυτά. Είναι λοιπόν σαφές ότι το θέμα δεν μπορούμε να το λύσουμε στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να επισημάνουμε τα προβλήματα και να καλέσουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους να αναζητήσουν λύσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, θα τα καταφέρουμε τελικά όλοι μαζί καλύτερα από ό,τι τα κατάφερα εγώ μόνος μου στο σχέδιό μου γιατί εντωμεταξύ μου κατατέθηκε ένα σχέδιο από την Freeport και από την ETF. Ε Έτσι λοιπόν, αν ε, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν κάποια λύση, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρξει και μια συγκεκριμένη διατύπωση για τους λιμένες. Όσον αφορά τώρα στην αυτονομία των λιμένων, αυτό είναι κάτι που δεν ικανοποιεί όλους, κυρίως τους συναδέλφους που έρχονται από την Ισπανία. Όταν όμως πρόκειται για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, ε, κατά την άποψή μου, τα λιμάνια, οι λιμένες ε, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το κόστος ως εργαλείο και όχι να δέχονται, να εξαναγκάζονται σε λύσεις από τις κρατικές κυβερνήσεις. Υπάρχουν σε κάποιες χώρες κάποιες ε, μέσες λύσεις, χρησιμοποιείται ο μέσος όρος ε, για δαπάνες και μετά το κόστος αυτό επεκτείνεται σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Αν αυτό ισχύει, τότε αυτό ε, κατά την άποψή μου αντιβαίνει ουσιαστικά στο πνεύμα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Γιατί αν θέλετε αυτό είναι μια οριζόντια επιδότηση. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των, των σκιωδών και κατανοώ κάποιους ε, που πιστεύουν ότι αυτά όλα θα δημιουργήσουν ε, προβλήματα στις πατρίδες τους αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε ακόμα και αν γνωρίζω ότι το Συμβούλιο δεν ε, θα ανταποκριθεί ιδιαίτερα. Τελευταίο θέμα, οι διαβουλεύσεις με τους χρήστες και εποπτεία και για τα δύο θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια λύση που να ταιριάζει τα πάντα και να βολεύει όλους. Οι διαβολεύσεις με τους χρήστες έχει νόημα μόνο εάν οι χρήστες είναι ενημερωμένοι για τον καθορισμό της αποζημίωσης ο τρόπος και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις, αυτό είναι θέμα των λιμανιών. Και στην εποπτεία το βασικότερο είναι να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας Υπάρχει βέβαια αυτό σε αρκετές ε, χώρες. Τώρα κατά πόσον ε, θα είναι ένα δικαστήριο ή ε, μια άλλη υπηρεσία καρτέλ, αυτό θα κρίνεται στην κάθε μία χώρα. Τώρα, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους και αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Τα έχουμε ήδη θίξει ακροθυγώς της Ενδριάσεως των σχεδόν Και αναφέρομαι στο εξής, το κατά πόσον θα πρέπει να εξαιρετούν οι μικροί λιμένες γιατί ενδέχεται η γραφειοκρατία να διονγκωθεί και τα μικρά λιμάνια ε, ενδέχεται να μην επωφεληθούν από τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αυτά καλό να τα σκεφτούμε σοβαρά όμως δεν θα πρέπει να έχουμε κατά νου μόνο την εμπορευματική κίνηση γιατί ε, στις περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν και τα λιμάνια με μεγάλη κίνηση επιβατών. Άρα δηλαδή το όλο θέμα είναι κάπως σαφές και πρέπει να το δούμε. Κάτι άλλο τώρα. Ποιος ορίζει ποια οργανωτική μορφή θα έχουν οι λιμένες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, Managing Authority ή αρμόδια αρχή. Νομίζω ότι τα ίδια τα κρατημέλη έχουν εδώ ε, τον τελικό λόγο, ο κύριος Βαντάλ κατέθεσε αυτή την πρόταση. Και όσον αφορά τώρα τον περιορισμό των προσφερόντων υπάρχει κάποια συζήτηση. Μερικοί προσφέροντες, οι μπίντεροι γνωστοί, η διατύπωση για αυτούς είναι πάρα πολύ ευρεία και ίσως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση να περάσουμε από έναν κλειστό σε έναν ανοιχτό κατάλογο. Αλλά πρέπει να το δούμε και να δούμε και, τις, ε, και τη διατύπωση και τις λεπτομέρειες. Τελευταία μου παρατήρηση, οι ε, που έχουν πολύ κυρίως όσον αφορά στη T-Port αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός αν δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι λιμένες. Αυτό δεν αφορά την εμπορευματική κίνηση, τα φορτία, γιατί τα φορτία εξαιρούνται έτσι κι αλλιώς, αφορά κάτι άλλο στο μέλλον, θα πρέπει όμως να το δούμε γιατί πιστεύω ότι αυτή την αντίφαση και τη σύγκρουση θέλουμε να την αποφύγουμε όλοι μας, που ναι μεν τώρα είναι θεωρητική αλλά στο μέλλον μπορεί να γίνει ε, πραγματική. 9-10 Νοεμβρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Θέλω επίσης να πιστεύω, επειδή αυτό είναι to be confirmed, αυτό θα αποφασιστεί στη συνεδρίαση των ε, σκιωδών εισηγητών. Και θα δούμε και ποια θα είναι η πρότασή μας σχετικά με το θέμα των επιδοτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Βόζεμπερκ, παρακαλώ. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο εισηγητή. Έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Δεν ήταν εύκολο κείμενο, δεν είναι εύκολο κείμενο αυτό που έχουμε ενώπιόν μας. Ε, έγινε και αντικείμενο μιας πορείας συμβιβασμού. Είναι μια καλή βάση για συμβιβασμό αυτό το κείμενο. Στις συζητήσεις και στις συναντήσεις που έχουμε κάνει στα πλαίσια των ε, σκιωδών εισηγητών. Έχει μπει ως βάση αυτό. Παρά τα αυτά χρειάζονται κάποια σημεία τα οποία θέλουν βελτίωση, αλλά και κάποια θα πρέπει να μετριάσουμε τη διατύπωση σε μερικές διατάξεις, οι οποίες όμως δεν είναι από τις βασικές που περιλαμβάνονται στο κείμενο. Δεν αποτελούν δηλαδή την, την ουσία του κανονισμού. Αρχικά σχετικά με κάποιες τροπολογίες για τα δικαιώματα των εργαζομένων που αναφέρονται τόσο στο πεδίο εφαρμογής συγκεκριμένα στην παράγραφο βα, όσο και στα άρθρα 4, 8, 10, 10α και σε άλλα σημεία εκφράζουμε συγκεκριμένες επιφυλάξεις διότι τέτοια θέματα δεν έχουν περιληφθεί στον κανονισμό διότι συζητούνται στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα θέματα αυτά να τα ρυθμίσει καθοριστικά από την αρχή μέχρι το τέλος ο κοινωνικός διάλογος. Ε, τα εργασιακά δικαιώματα επίσης ε, ξέρουμε ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εδώ ε, είμαστε μπροστά στην αρχή της επικουρικότητας. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται πολύ το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ενώ περιερίζεται σε άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τη λειτουργία των λιμένων. Αναφορικά με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον κανονισμό, πιστεύουμε ότι για να υπάρξει περισσότερη διευκρίνηση και σαφήνεια στο κείμενο, να μην υπάρχουν ε, ερωτηματικά και τόση αμφισβητήσεις, θα ήταν καλό να προσθέσουμε τον ορισμό της αρμόδιας αρχής. Σε σχέση τώρα με το άρθρο 3, που καταρχήν ήταν ένα σημείο έντονης αντιπαράθεσης και επιθυμούσε τη διαγραφή του ο κύριος Συγητής, καταφέραμε να βρούμε ένα συμβιβασμό στον οποίο περιγράφεται η οργάνωση του λιμενικού συστήματος της Ένωσης. Επίσης, σχετικά με το άρθρο 4, στην παράγραφο 4, θεωρούμε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του διαχειριστικού φορέα του Λιμένα η εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης στην εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή βάση για συμβιβασμό η τροπολογία 366 η οποία κάνει λόγο για το πώς εξασφαλίζεται η επαρκής πρόσβαση στις πληροφορίες. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Ε, σχετικά τώρα με τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων, πιστεύουμε ότι στο άρθρο 6 ο εισηγητής στο κείμενο που μας έχει εμφανίσει κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς προτείνεται μια νέα παράγραφος, η 3α, στην οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνει την υφιστάμενη νομολογία λέγοντας ότι η διαδικασία πρέπει να είναι διαφανής και χωρίς διακρίσεις. Παρά τα αυτά η εμπειρία μας δείχνει ότι η νομολογία πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα γιατί έχει και μία και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Έχει πολλές ερμηνείες και που θα μπορούσαν να, να οδηγήσουν σε νομικά διέξοδα, βεβαιότητες. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ενταχθούν στο συμβιβασμό κάποιες από τις τροπολογίες μας που περιγράφουν τη διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων. Είναι δηλαδή λεπτομερής η περιγραφή για να μην καταλείπονται αμφισβητήσεις ως προς αυτό που θέλουμε να διατυπώσουμε. Για να δώσουμε μεγαλύτερη σταθερότητα για τους επενδυτές στους οποίους κατατείνει η διευκρίνηση να είναι ε, απολύτως ξεκάθαρο το τοπίο της νομικής κατεύθυνσης. Στο άρθρο 8, σχετικά με τις τροπολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6, είμαστε της άποψη ότι οι εργασιακές κινητοποίησεις θα πρέπει να εξετάζονται ως επιλογή όταν έχει τελειώσει το πεδίο του διαλόγου. Δηλαδή οι κινητοποιήσεις το γνωρίζουμε όλοι ότι όταν ο διάλογος είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ανατραπεί ε, η προσπάθεια ή δεν έχει φτάσει στο να επιχειρηθεί, ε, παρακολεί τις εργασίες με, με κίνδυνο να έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές την πάυση της λειτουργίας του λιμένα και η παρακόλληση άλλων ε, λιμενικών υπηρεσιών που επηρεάζουν τους χρήστες του λιμένα και τις δραστηριότητες. Γι' αυτό εμείς λέμε ας πούμε ότι να εξαντληθεί ο, ο διάλογος πάντοτε βέβαια σε σεβασμό με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών όπου τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζονται. Στο άρθρο 10 πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που γίνεται αναφορά στο σεβασμό της εθνικής εργασιακής νομοθεσίας των κρατών μελών η αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις περιτεύει. Δεν θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει να εξαλειφθεί. Επιπλέον, στην παράγραφο 10α, νέα που προτείνεται στην εισήγηση, συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι εργάτες δέχονται την κατάλληλη κατάρτιση, καθώς και οι νέες δεξιότητες τους επιτρέπουν να έχουν μεγαλύτερες και καλύτερες, αξιότερες δηλαδή επιδόσεις, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της εταιρεία. Θεωρούμε παρά τα αυτά ότι στην παράγραφο 3 του νέου 10α δεν πρέπει να είναι τα κράτη-μέλη υπεύθυνα να αναπτύξουν μοντέλα που εξασφαλίζουν τις ε, διακυμάνσεις στη ζήτηση, αλλά η κοινωνική εταίρη. Επίσης, στο άρθρο 12 θέλουμε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζεται ο κανονισμός σε θαλάσσιους λιμένες του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου προκειμένου να αποφεύγεται και ο διοικητικό ο διοικητικός φόρτος <laughs> ναι, να συντομεύσω μέσω τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Και το κόστο για του λόγω λιμένε. Αναφέρω τι τροπολογίε αριθμητικά μόνο, την 566 από το ECR, την κοινή 566 με τους, 565, ε, 566 με του συναδέλφου και την τροπολογία 567 του συναδέλφου του κυρίου Κύρκου από το, ε, την ομάδα των Σοσιαλιστών. Αντίστοιχη θέση έχουμε και για του θαλάσσιου λιμένε του συνολικού διευρωπαϊκού δικτύου. Αναφορικά τέλο με τα τέλη των λιμανικών υποδομών στο 14 παράγραφο 4 Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ρητή αναφορά ότι τα τέλη λιμενικών υποδομών μπορούν να διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις εμπορικές πρακτικές που σχετίζονται σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών, όπως περιγράφουμε στο 594. Και τελειώνω οριστικά, κύριε Πρόεδρε, με, σχετικά με τις τροπολογίες για την ανεξάρτητη εποπτεία. Πιστεύουμε ότι περισσότερες από αυτές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και επίση το κείμενο που μας έχει παρουσιάσει ο κ. Συγητή, υποστηρίζει μια διοικητική απλούστευση ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφανίζουν ένα μηχανισμό διαχείρισης των καταγγελιών ούτω ώστε να συγκεντρώνονται και να μπορούν να ελέγχονται καθοριστικά. Σα ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη αν πήρα λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω όμω, ε, μόνο να σα υπενθυμίσω ότι δεν τις ξέρουν όλοι τις λεπτομέρειες των τροπολογιών. Κανονικά κάνει κανείς μία σύνοψη και το πρόσεξα και σε άλλες εκθέσει, ε, σε άλλη περίπτωση και άλλοι είπαν πράγματα που δεν τα ήξεραν οι υπόλοιποι. Τέλο πάντων δεν πειράζει, ο κύριο Πέτερ Φαντάλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του θέματος και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή που έχει υιοθετήσει μια επικοδομητική προσέγγιση. Το εκτιμούμε αυτό. Ωστόσο, δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα και τα προβλήματα και πέντε από αυτά είναι τα πιο σημαντικά για εμάς. Πρώτα απ' όλα ο εισηγητής ε, ο ίδιος έχει πει ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε 9 και 10 Νοεμβρίου στην Επιτροπή, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να βιαστούμε. Καλύτερα να πάρουμε λίγο περισσότερο χρόνο αν χρειάζεται, ε, ένα μήνα, δύο μήνες, ε, όπως έχει συζητηθεί και στο παρελθόν. Είναι καλύτερα να είμαστε σχολαστικοί παρά να βιαστούμε ε, ει βάρο της ποιότητα και να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέτρα που δεν του ταιριάζουν. Μετά, είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη λιμένων στα διάφορα κράτη-μέλη με διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά τον τρόπο λειτουργία τους. Γι' αυτό εμείς θα θέλαμε να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευχέρεια τα κράτη-μέλη να επιλέγουν τους τρόπους που αυτά θα λειτουργούν. Δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε ε, τα πάντα στις Βρυξέλλες να αποφασίζονται. Τρίτον, κάτι που πιστεύω ότι θα δημιουργήσει ε, συζητήσεις ε, θα συνεχιστούν οι ενδιαφέρουσε συζητήσει πάνω στο θέμα αυτό είναι το θέμα των κοινωνικών εταίρων. Κατά την άποψή μου, ε, τα κράτη-μέλη έχουν οργανώσει τον δομημένο κοινωνικό διάλογο ε, επί σειρά ετών και λειτουργεί πολύ καλά, επομένω όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα θα πρέπει να επαφίονται σε αυτόν. Τέταρτον, όσον αφορά την διαφάνεια, δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου να υπάρχουν κρυφές πληρωμές, οι ροδοκίες και η μέρημνά μας θα πρέπει να είναι να μην υπάρχει καθόλου στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ε, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν και όλοι οι σκιώδεις, θα έλεγα, σε αυτό το ζήτημα, το ζήτημα της διαφάνειας. Πέμπτο. Κοιτώ την συμβιβαστική 17 όπου αναφέρεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ε, εποπτικής αρχής. Αυτό, κατά την άποψή μας, δεν είναι επιθυμητό, γιατί δημιουργεί μεγάλο διαχειριστικό άχθος και ε, υπερβολική νομοθεσία για ένα ζήτημα που δεν χρειάζεται. Αυτά είναι τα πέντε ζητήματα που για το ECR είναι τα πλέον σημαντικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σα πω ότι οι συζητήσει προχωρούν ικανοποιητικά. Ευχαριστώ. Φυσικά το τελικό κριτήριο είναι πάντα η ποιότητα, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε μόνοι μα τη δουλειά μας. Η κυρία Γκεσίνε Μάισνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Φλέκενστάιν, τον εισηγητή, για την μέχρι τώρα δουλειά του. Ε, πραγματικά πρέπει να το πω. Προχωρήσαμε, προχωρήσαμε αρκετά. Και ισχύει το εξή, ότι το σχέδιο τη έκθεση ε, σε, σε πολλού από εμά ε, δεν μα άρεσε, γιατί ήταν τελείω διαφορετική από την πρόταση Κομισιόν. Η Κομισιόν είχε πει η αγορά να είναι στο επίκεντρο. Ο εισηγητή ε, προσέθεσε πολλά κοινωνικά στοιχεία και είπε ότι τον ανταγωνισμό δεν τον χρειαζόμαστε απαραίτητα γιατί έτσι κι αλλιώ ήδη υπάρχει. Καταλήξαμε λοιπόν σε συμβασμό που κατά την άποψή μου ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και αυτό κατέστη σαφέ και από τι μέχρι τώρα παρεμβάσει. Ε, θα ξανασυναντηθούμε αυτή την εβδομάδα και ένα βασικό σημείο είναι το κοινωνικό σκέλος. Αυτό το έφτιαξαν όλοι. Πράγματι είναι αλήθεια ότι η ε, το κοινωνικό στοιχείο έχει σχέση και με την επικουρικότητα, άρα και με τα κράτη-μέλη και κατανοώ βεβαίως ότι θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες εργασίας ε, στους λιμένες. Αν όμως ε, το Φεβρουάριο υπάρξει μια καλή πρόταση όπως έχει ανακοινώσει ο εισηγητής γιατί άκουσα ότι κάτι ψήνεται. Ε, αν λοιπόν ε, συμφωνήσουμε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αυτή την οδηγία για τους εργαζόμενους τους λιμένες δεν μπορούμε να την εκλαμβάνουμε ως δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι στρατηγική. Ε, τι θα κάνουμε με τα μεγάλα ε, σκάφη, τα εμπορικά. Ίσως ε, λοιπόν ε, να περιμένουμε καταρχήν αυτή την πρόταση. Και αυτό που ήδη βρίσκω καλό είναι το πεδίο εφαρμογής. Νομίζω πολύ σωστά συμφωνήσαμε ότι το πεδίο εφαρμογής είναι αρκετά εκτεταμένο, καλό είναι αυτό. Η διαφάνεια της αποζημίωσης είναι σωστή η πρόσβαση στην αγορά και αυτό είναι ικανοποιητικό και αυτό προέκυψε από το συμβασμό για μένα και το έχω ήδη πει το βασικότερο είναι ότι τα λιμάνια στα κράτη-μέλη είναι τελείως διαφορετικά και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε τώρα να επιβάλλουμε κάτι το οποίο αμφισβητεί το ήδη ισχύον. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό και νομίζω ότι προχωράμε πολύ καλά με τους ε, συμβασμούς. Πάμε τώρα σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι τα ιδιωτικοί λιμένες. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικοί λιμένες όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στη Γερμανία. Λίγοι αλλά υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα λιμάνια ε, όταν θα προσφέρουν υπηρεσίες προφανώς θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή ε, της οδηγίας. Γιατί είναι σαφές όταν μου ανήκει κάτι και θέλω κάτι να κάνω δεν μπορώ να μου πει ο άλλος πώς θα το κάνω. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για τους ε, συμβασμούς Pilot Exemption Certificates αυτή ήταν μια τροπολογία των φιλελευθέρων οι ε, καπετάνοι που είναι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να έχουν πρόβλημα ε, όταν γνωρίζουμε καλά το λιμάνι. Ας πούμε η Αμβέρσα είναι ένα λιμάνι όπου υπάρχουν ε, τελείως διαφορετικές ε, ρυθμίσεις για τους οδηγούς από ό,τι σε άλλους λιμένες. Βεβαίως θα ήταν καλό κάπου τον Νοέμβρη να τελειώνουμε, γιατί οι περισσότεροι στους λιμένες επιθυμούν να, έχουν μια συγκεκριμένη λύση. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πιεστούμε τόσο πολύ ε, και να καταλήξουμε σε κάτι το μεσοβέζικο, ε, θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, γιατί υπήρξαν τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την αποζημίωση, ε, για μένα υπάρχει το ισπανικό μοντέλο και κάθομαι και δίπλα σε μια Ισπανίδα είναι ένα μοντέλο του μέσου όρου. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε όλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπω και ένας κύριος άλλος από την Ισπανία με κοιτάει. Μπας περιπτώσει εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση που να ικανοποιεί όλους. Ο κύριος Τέλιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλή ανάρρωση. Well, thank you very much, Chair, and I've missed... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου λείψατε. Αλήθεια σας λέω. έκανα εγχείρηση στο γόνατο και τώρα το καινούργια μου κλείδωση θα τη πάρει λίγο καιρό να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Έρχομαι στο θέμα των λιμένων. Ποτέ δεν το ξέχασα καθόλου τη διάρκεια της ε, ανάρρωσης μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φλεκενστάιν για την εξαιρετική εντυπωσιακή δουλειά που έχει κάνει ως εισηγητή για το θέμα αυτό. Δυστυχώ τα αποτελέσματα αυτού του εξαιρετικού έργου έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού και καταδεικνύουν ορισμένα τα πολύ πιεστικά προβλήματα που συνεχίζει να έχει ο κλάδος. Οι ειδικοί επιθυμούν μεγαλύτερη σαφήνεια, να είναι πολύ πιο ξεκάθαροι οι κανόνες όσον αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. Και αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και επενδύσεις στον τομέα αυτών. Το κείμενο όσο έχει αυτή τη στιγμή πολύ λίγο συνεισφέρει σε αυτήν την σαφήνεια, πολύ λίγο ξεκαθαρίζει αυτούς τους κανόνες για τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Ενώ ταυτόχρονα η Επιτροπή ανακοινώνει μάλλον απειλή ότι πρόκειται να κινήσει διαδικασίες εναντίον κρατών μελών για παραβιάσει των κανονισμών για τι κρατικέ ενισχύσει. Θα δούμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλο του, του έτου. Λυπάμαι, δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επίπεδο που θα έπρεπε. Η πολιτική μου ομάδα θεωρεί ότι ακριβώς επειδή θα διονυστεί αυτή η ανασφάλεια δικαίου, θα ήταν καλύτερα να είχαμε υιοθετήσει ε, την μέθοδο της οδηγίας, δηλαδή να ήταν οδηγία αυτή η νομοθεσία και όχι κανονισμός. Βεβαίως, όπως είναι φυσικό, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε επικοδομητικά και να φροντίσουμε έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα αυτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ομάδα μου θα ήθελε να υιοθετηθούν οι εξαιρεσει πριν να ολοκληρωθεί η συζήτηση και το έργο πάνω στο PSR, πάνω στην, στον κανονισμό αυτόν. Έχω ακούσει από πολλού να μου λένε ότι αυτή η νομοθεσία δεν είναι επαρκής, δεν είναι καλή. Γι' αυτό και εμείς η πρώτη τροπολογία που υποβάλαμε ε, ήταν να, να την καταψηφίσουμε στο σύνολό τη, να, μην ε, υιοθετηθεί ε, ο κανονισμός για τις υπηρεσίες λιμένων. Γιατί έχουμε κάνει τόσες πολλά πισωγυρίσματα και τόσο πολλά μπροσπίσω μάλλον και τόσο πολύ δεν είναι ξεκάθαρες μια σειρά από λεπτομέρειες που νομίζω κανείς δεν αντιλαμβάνεται ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας. Συμφωνώ και με την κύριο Φλέκενστάιν. Ως προς το εξή, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος ενός ε, λιμένα. Ένας μικρός, ένα μικρό λιμάνι στα, στην Αγγλία. Για παράδειγμα ένα λιμάνι όπως η Οστάνδη. Είναι ένα λιμάνι στο οποίο δεν γίνεται ε, δεν έχει μεγάλη εμπορική κίνηση. Πρέπει να έχει διαφορετικού κανόνες από ένα μεγαλύτερο εμπορικό. Αλλά και πάλι, το μέγεθος της εμπορική κίνησης δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιούμε. Ένα άλλο κριτήριο, για παράδειγμα, σημαντικό είναι πόσο χρησιμοποιείται από ferry boat το λιμάνι. Επομένως, χαίρομαι που κάναμε αυτή τη ζήτηση και που έχουμε προοδεύσει μέχρι τώρα, αλλά θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο μπροστά. Μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να ήμασταν σε πολύ καλύτερο σημείο από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι σκιώδη ηγητέ, αλλά επειδή ζήτησαν πάρα πολύ το λόγο, ε, θα περιορίσουμε το χρόνο αγόρευση σε δύο λεπτά. Ντομινίκ Κρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φλίκενστάιν για το πολύ περίπλοκο έργο που πετέλεσε. Κάτι καινοφανέ το θέμα τη προόδου, τη προβληματισμού κλπ. Υποδειγματική δουλειά. Και είναι αναγκαίο διότι αν γίνεται όπως εάν ε, ε, δεν λειτουργεί όπως είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν έχει η απόπειρα σε αρισμένα αθλήματα απορρίπτεται κανείς, αποκλείεται λοιπόν δεν θέλω να επανέλθω στα όσα ήδη υπόθηκαν το πρώτο ερώτημα που θα θέσω αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επέκταση λοιπόν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας στο κεφάλαιο 1 Τροπολογία 1βα. Εκεί που διευρύνεται αρκετά σημαντικά το πεδίο εφαρμογή και το θέμα. Που είναι αρκετά περιορισμένο κανονικά. Αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα κανονιστικό. Μπορούμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή. Ή αντιθέτω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Και αλλάζοντα τον ορισμό, αλλάζουμε τον αντίκτυπο που έχει η οδηγία ή ο κανονισμό. Το λέω αυτό διότι κάποιοι συνάδελφοι πριν από μένα έκαναν αυτό το σχόλιο ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια προβλήματα αυτή η προσέγγιση όπως τα κοινωνικά θέματα ή ε, περιβαλλοντικές πτυχές του κώδικα εργασίας. Η περιβαλλοντικες πτυχες του κωδικα Επιτροπή θα μας πει πρέπει να τηρήσουμε τα πλαίσια του κανονισμού όπως το θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι πρόκειται για την, το δικαίωμα πρωτοβουλίας. αν επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής παρεμβαίνουμε στο δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Και μετά δύο παρατηρήσει συντομία. Όπω υπόθηκε, θα πρέπει να αποκλείσουμε τα μικρά λιμάνια ή ε, αυτά τα πολύ απόμακρα που λόγω, για λόγους γεωγραφικούς και για λόγους εφαρμογής και προσέγγισης για το διεθνή ε, ανταγωνισμό χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. θα σταματήσουμε, σε ποια κλίμακα, πώς θα θέσουμε το όριο είναι θέμα, το πρόβλημα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος να τις επενδύσεις. Αυτό είναι ε, αντιπαραγωγικό. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί και να ελοποιηθεί, δημιουργούνται προβλήματα εμπιστευτικότητα. Αυτό το σημείο λοιπόν θα ήμουν ικανοποιημένο αν θα μπορούσαμε τελικά να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Βονταλού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Κνούτ Φλέκενστάιν για την έκθεσή του και για τη δουλειά που έκανε. Που δεν ολοκληρώθηκε άλλωστε. Δεν τελείωσε. Είναι σημαντικότατο το σημείο αυτό. Η έκθεση άλλαξε σημαντικά την, την φιλελεύθερη προσέγγιση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το χαιρετίζουμε αυτό. Αφήνει περιθέριο λιγμών στις αρμόδιες αρχές έτσι να παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες και να γίνονται σεβαστές περιβαλλοντικές πτυχές και κοινωνικές πτυχές και συνέχιση παροχή των υπηρεσιών. Κάτι άλλο να υπογραμμίσω. Ξέρω ότι συνεχίζονται συζητήσει επ' αυτού. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να αποκλείσουμε όπως τις υπηρεσίες ε, πλοήγησης και ε, της ε, ρημούλκησης που αφορούν, δεν είναι εμπορικέ υπηρεσίες, αλλά ασφαλείας. Αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων, των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα δεν θα πρέπει να έχουμε διαφοροποιημένο διαφοροποιημένη προσέγγιση αυτή τη υπηρεσία για να μην πειράσουμε την ασφάλεια των ε, λιμένων και την ασφάλεια των εργαζομένων. Να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε κάποιων κρατών μελών που επιβάλλουν σε εκείνον που ασκεί τη ρημούλκηση υποχρέωση σημαία ε, που φέρει το σκάφος και αριθμό ε, ναυτικών. Ε, δεν θα πρέπει... Δεν πρέπει να διευκολύνουμε να μπουν νέοι πάροχοι που θα χρησιμοποιούν σημαία ευκαιρία και θα υπονομεύουν την ποιότητα τη απασχόληση, κοινωνικέ πτυχέ και την ασφάλεια των λιμένων. Θα έπρεπε να έχουμε συμβιβασμό, να δώσουμε δυνατότητα στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να εξαιρέσουν αυτού του είδου τι υπηρεσίε θα έπρεπε να έχουμε σαφή ορισμό της αρμόδιας αρχής. Θα πρέπει και έχουμε ένα κείμενο που δεν ε, αναφέρει τα βασικά σημεία του κανονισμού. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στον αφορά τους ορισμούς. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Έκλεισε τώρα ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, τελευταία ομιλήτρια, παρακαλώ. Ε, κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ήταν δύσκολο το έργο του. Ο εισηγητής είχε δύσκολο έργο. time because Λοιπόν, κάτι που είπα και προηγουμένω. Εν γέννη υπήρξε κάποια πρόοδο. Υποστηρίζουμε ορφανώς τροπολογίε που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να εξαιρέσουν τα μικρά λιμάνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και τροπολογίε στηρίζουμε που αφορούν τη διαφωνία τη χρηματοδότηση για του κρατικού λιμένε και συμμόρφωση και αυστηρού κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει και για κάποιες παρεκκλήσεις συμφωνούμε βλέποντας την εξαίρεση για την ανταγωνιστική αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά όμως που είναι κρεμή. Δεν υπήρξε επαρκής πρόοδος για μας όσον αφορά τη στάθμη των σκάφων, διαχείριση αποβλήτων, ρημούλκηση σκαφών κλπ και συμπερίληψη των πορών τροπολογιών για κοινωνικέ πτυχέ, κοινωνική προστασία και δικαιώματα ε, εργαζομένων και εργοδοτών και προστασία των εργαζομένων. Δεν θέλουμε να επανέλθουμε στο παλιό σχήμα που είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε ιδιωτικοποιημένα λιμάνια, εδώ και 20-30 χρόνια τώρα και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και δεν έχουμε προβλήματα με τη χωρητικότητα. Οπότε αυτό είναι σαφέστατο. Επίσης, είμαστε αντίθετοι στις τροπολογίες που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Φορέα που θα διευθυνθεί τις διαφορές, κάτι που έθεσαν συνάδελφοι. Επίσης, με εθνική αρμόδια αρχή σε όλα τα κάτι μέλη που θα πρέπει να ελέγχει τη συμμόρφωση. Δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Εν γέννη λοιπόν υπήρξε κάποια μετακίνηση. Υπέβαλα μόλις εννέα τροπολογίες. Εκτός αν υπάρχει κάποια σοβαρή μετακίνηση από όλες τις πλευρές όσον αφορά τα σημεία που έθιξα, δεν νομίζω ότι φορά μόνο εμένα και τον Εμένο Βασίλειο. Θα απορρίπταμε αν δεν υπάρχει λοιπόν επαρκής μετακίνηση την πρόταση. Παρόλη την πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, την πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει καταβάλει ο συγγητής. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά την άποψή μου, την οποία σας παρουσίασα και τον Ιούνιο, με εκπλήσει το γεγονό ότι συνεχίζουμε να συζητάμε έναν κανονισμό παρά το γνωρίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα μια αναθεώρηση της αξιολόγησης αντικτύπου όπως είχαμε ζητήσει και το οποίο θα ήταν και ε, συναφές με τις πρωτοβουλίες για το Better Regulation. Μιλάμε για μια βελτίωση του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας και είναι προφανές ότι θα έπρεπε αυτό να εξισορροπείται με μια βελτίωση των εργατικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών ε, θεμάτων. Επομένως εκπλήσωμαι που δεν αναφέρονται αυτά τα ζητήματα αρκετά. Ε, συμφωνώ με τη συνάδελφο Κριστίν για την σημασία που έχει η ασφάλεια στον κλάδο και η ποιότητα των διαθέσιμων ε, δουλειών στον κλάδο αυτό και ότι πρέπει να το προστατεύσουμε. Τον Ιούνιο είχαμε συζητήσει και είχαμε την εντύπωση ότι θα υπάρξουν και πρόνοιες οι οποίες θα διασφαλίζουν τα θέματα αυτά, τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα. Επομένω, δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα μπορέσουμε να πείσουμε του κοινωνικού εταίρου να υποστηρίξουν και να υιοθετήσουν και να αποδεχτούν αυτόν τον κανονισμό, εάν δεν συμπεριλάβουμε τέτοιε προβλέψει. Συμφωνώ επίση ε, και με άλλου συναδέλφου αλλά δεν συμφωνώ μάλλον με τις ε, απόψεις άλλων συναδέλφων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είμαστε όλοι σύμφωνοι οι προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και το βλέπω λυπηρό που κάποιοι από του υπουργού από το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν να τραβήξουν αυτόν τον κανονισμό προ μια άλλη κατεύθυνση. Διαπιστώνουμε και σε ορισμένε τροπολογίε από διάφορε ομάδε να προσπαθούν να διαγράψουν συγκεκριμένε προβλέψει του κανονισμού και αυτό ε, πιστεύω είναι απαράδεκτο γιατί έχουν γίνει προσπάθειες να βελτιωθούν τα διάφορα πρότυπα κυρίως εκείνα που αφορούν στην κατάρτιση. δεν είναι το ίδιο να αναφερόμαστε στην πρόσβαση στην πληροφορία με το να υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Αυτά μόνο μπορώ να σας πω μέσα στα δύο λεπτά που είχα. Ευχαριστώ. Ε, ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο που έκαναν ως τώρα διαπιστώνω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον κανονισμό αυτόν. Καταλαβαίνω τους Βρετανούς συναδελφούς αλλά υπήρξαν πολλοί, πολλές οδηγίες ε, για το θέμα των λιμένων που δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το άρθρο 6.3α το οποίο αντικαθιστά το 7. Έχω μια ερώτημα σε σχέση με αυτό. Τι σημαίνει και πώς σχετίζεται με την οδηγία για τις παραχωρήσεις. Οι παραχωρήσεις ε, επιτρέπονται ή απαγορεύονται με βάση το νέο άρθρο αυτό. Δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα των τελών που είναι πολιτικά ευαίσθητο. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Τα κράτη-μέλη θα ε, ε, ε, επιλέγουν ποια είναι τα τέλη ή η διαχειριστική αρχή του κάθε λιμένα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Μετά, άρθρα 15, 16 και 17. Εδώ διαπιστώνω ότι ο κύριος Φλέκενστάιν έχει απομακρυνθεί από τη θέση του Συμβουλίου και θα ήθελα να μας εξηγήσει γιατί το κάνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να επισημάνω το εξής. Ε, νομίζω ότι ο εισηγητής ε, μας κατησύχασε, εγώ τον γνωρίζω, είναι πολύ αποτελεσματικός ε, βουλευτής και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Γι' αυτό η δική μου πολιτική ομάδα θα τον στηρίξει. Οι ανησυχίες μας καλύφθηκαν και ο διάλογος που γίνεται τώρα ευελπιστώ ότι θα τελεσφορήσει. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να θυγούν, που δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφή. Ε, γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω πρώτα απ' όλα το εξή. Εμείς επιθυμούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ε, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων έχουν μεγάλη, έχει μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε θα απελευθερώσουμε όλα τα λιμάνια είτε πολύ σύντομα δεν θα έχουμε πια αυτή την ευκαιρία. Και υπάρχουν και ολόκληροι τομείς ε, όπου η αλυσίδα των μεταφορών πρέπει να παραμείνει άθικτη για τη βιομηχανία. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλες αυτές οι εξαιρέσεις. Και όσον αφορά τα τέλη λιμένων, ο εισηγητής ε, λέει ότι τα τέλευτα θα πρέπει να ορίζονται από τις αρμόδιες ε, επιτροπές. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Ισπανία λόγω του συντάγματός μας. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτό που σας είπα και διαφωνούμε. Πρέπει εμείς ε, να μπορούμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική λιμένων ε, που θα καθορίζεται από τη διαφάνεια. Ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Σημαντικό, όπως σας είπα, τα τέλη των λιμένων να είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων. Άρα δηλαδή αυτό που παίζει ρόλο είναι να γίνεται γενικά συζήτηση για τις ε, υπηρεσίες που παρέχονται από τους λιμένες. Τελειώντας λοιπόν θέλω να πω ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους ε, επιβάτες ε, θα προσφέρονται ελεύθερα. Μιλάω βέβαια πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά είχα να σας πω. Ακούσαμε τις διάφορες παρεμβάσεις Υπάρχουν κάποια θέματα που μας ενδιαφέρουν, μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και όπως σας είπα είμαι πεπισμένος ότι ο διάλογος θα είναι θετικός και εμείς επιθυμούμε να μεριμνήσουν όλοι για να τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μάρη Κριστίνα Νοτού, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγκρίνω το κείμενο του 2013 της Επιτροπής με το κείμενο που έχουμε σήμερα μπροστά μας και διαπιστώνω το με ευχαρίστηση ότι κινηθήκαμε προς τη συστή κατεύθυνση εξέλιξης. Ήταν θετικές. Από το 2015 αναγκάστηκε η Επιτροπή να αναθεωρήσει τις απόψεις της και ε, να μετριάσει την προσπάθειά της να φιλελευθερωποιήσει, ε, να απελευθερώσει μάλλον την αγορά για ζητήματα όπως το dredging ή τη, τη ρημούλκηση ή την πρόσδεση σε προβλήτες. Το 2014 το Συμβούλιο έχει επίσης εξα, ε, ε, ορισμένες από τις υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό Και επίσης διαπιστώνουμε ευχαρίστηση ότι έχει αυξηθεί το μέρος ε, της ευθύνης που θα έχουν τα κράτη-μέλη, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα εκείνα να ρυθμίζουν την αγορά αυτή αν το θεωρούν ε, σωστό. Κάτι το οποίο θα ε, διευκολύνει κυρίως τα μικρά λιμάνια. Αυτά ήταν θετικά. Ωστόσο, στα ζητήματα των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο μακριά γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένε προβλέψεις οι οποίες ε, προέρχονται από την Επιτροπή. Θα ήθελα να προτείνω τη διαγραφή της ετελεγικής σκέψης 5, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 165 της ε, συνθήκης και το οποίο αναφέρεται στην εξέλιξη των περιορισμών στην ε, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ε, θέμα στο οποίο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, όπως αυτό έχει πολλές φορές διατυπωθεί, από το 2005 κατά τη διάρκεια της συζητήσεων για το σχετικό άρθρο της συνθήκης. Επίσης, η αποχρέωση των αρχών διαχειριστικών των, λιμάν, των λιμένων να αποστέλουν στην Επιτροπή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα πιστεύω ότι θα πρέπει να διαγραφεί γιατί δεν θα θέλαμε μέσω αυτή τη διαδικασία να μπορεί η Επιτροπή να λάβει πληροφορίε που θα τη δώσουν την δυνατότητα να λάβει μέτρα στο υπερεθνικό επίπεδο εναντίον των συμφερόντων των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ομάδα μου, του NGL, Ευχαριστώ τον Κνούτ Φλέκενστάιν για τη δουλειά που έκανα. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Εγώ είδα ότι γίνονται πολλές συζητήσεις. Με προβληματίζει το άρθρο 3 που έχει σαν στόχο να δώσει στις αρχές πολύ εκτεταμένες εξουσίες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, στο άρθρο 9 του κανονισμού λέει ότι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν για την παροχή των υπηρεσιών τους, για τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Προσωπική μου επιθυμία θα ήταν αυτό να μην αφορά τη διαχείριση των εμπορευμάτων στο μέλλον. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ελευθερία που χορηγείται στις λιμενικές αρχές μήπως δημιουργήσει την κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση των διαφόρων φορέων. Δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο. Αυτό αφορά και τα μικρομεσαία λιμάνια αλλά και τα μεγάλα λιμάνια. Όλα τα λιμάνια δεν έχουν τον ίδιο αριθμό παρόχων υπηρεσιών ή παρόμοιο αριθμό, άρα πρέπει να φροντίσουμε όλοι να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκύρκος, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον συνάδελφο Φλακενστάιν για την εξαίρετη δουλειά που κάνει σε ένα τομέα που συναντάει μεγάλε αντιστάσει. Εκτιμώ ότι η πρότασή του βελτιώνει στο ορισμένα σημεία την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η θέσπιση πλαισίου για τι λιμενικέ υπηρεσίε παραμένει αναγκαία για τη δημιουργία διαφανού και νομικά σταθερού περιβάλλοντο, που θα ευνοήσει τη λιμενική δραστηριότητα. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο θέματα που έφεξε ο κύριο Το ένα είναι τα μικρά λιμάνια, αυτά που έχουν μικρή οικονομική δραστηριότητα, οπότε η αύξηση, η παράλογη αύξηση των διοικητικών δραστηριοτήτων θα τους δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Άρα πρέπει να τηρηθεί η διαφάνεια, αλλά να έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση για το τι πρέπει να κρατάνε. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι οι λιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να προστατεύονται έναντι λιμένων που δεν ε, προστατεύονται, που δεν υπόκειται στα ίδια κριτήρια οργάνωσης και λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και τέτοια έχουμε εμείς στην ανατολική και την νότια πλευρά της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φλέγκενστάιν για όλη τη δουλειά που έκανε. Να του πω ότι Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια ταχύτερο δυνατόν, διότι αντίθετα το πακέτο των σιδηροδρόμων που όλο και επιταχύνουμε, εδώ όλο επιβραδύνουμε. Και είναι τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προχωρήσουμε. Να επαναλάβω για την εξαίρεση των υπηρεσιών πλοήγησης. Ε, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά διότι οι καπετάνοι των πλοίων μπορούν να είναι καλοί και άγιοι και υπέροχοι, αλλά ένα από αυτά που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι γίνονται λιγότεροι έλεγχοι από την παλιά. Και έχουμε πλοιάρχους που δρούν σαν πιλότοι ε, στην κίνησή τους στο λιμάνι και αυτό δεν θέλουμε να το δούμε. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουν. Θα πρέπει λοιπόν οι πλοηγοί, οι πιλότοι να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ε, τα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τις κριτικές ενισχύσεις. Αυτό δεν το συζητούμε μόνο στον τομέα των μεταφορών. Είναι ένα θέμα που ξεπερνά τον τομέα των μεταφορών, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μετά για τα ισπανικά λιμάνια, όπως αναφέρθηκε, αυτό είναι κάτι που συνδέεται με το Σύνταγμα. Το Ισπανικό Κοινοβούλιο αποφασίζει για τα τέλη τα λιμενικά μετά από πρώτερες συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Ελπίζουμε αυτό τελικά να γίνει κατανοητό και αντιληπτό. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε καταρχάς την ποιότητα της διεξαχθής σας συζήτησης, ε, την ποιότητα των υποβληθισών τροπολογιών και την ποιότητα της εκθέσεως του κυρίου Φλέκενστάιν. Η έκθεση βασίζεται στις πιο πρόσφατες ε, κυκλοφορούσες ιδέες και ο χρονισμός είναι σημαντικότατος. Στο ψήφισμά σας για τη Λευκή Βίβλο παραδεχθήκατε τον, τη σημασία που έχει ο κανονισμός και τη σημασία προόδου της προτάσεως και μετά από την ανάγνωση του Συμβούλιο η επόμενη Προεδρία, η Ολλανδική, επιθυμεί διακαώς να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μαζί σας, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερο πλαίσιο για τους λιμένες μας. Είναι κρισίμου σημασία οι λιμένες όχι μόνο για την αλυσίδα της κινητικότητας, αλλά και για τις επενδύσεις που μπορούν να προσελκύσουν. Για τις τροπολογίες δεν θα ήταν πολύ σόφρον ή ενδιδεγμένο σε αυτή τη φάση να επισέθω σε λεπτομέρειες σχολιάζων κάποιες από τις τροπολογίες. Θα περιοριστώ σε κάποιες αντιδράσεις. Όσον αφορά τα κεφάλαια 3 και 4, ε, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που βελτιώνουν σημαντικά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοστική διαφάνεια, για την αυτονομία των λιμένων, για το υποπτικό καθεστώς κλπ. Για τα τέλη επίσης και το καθεστώς των τελών, όπως ανέφεραν και κάποιοι, όπως η κυρία Μάισνερ, πιθανότατα εκεί υπάρχει κάποια λύση για να εξασφαλίσουμε σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας απόφασης των λιμένων, να μπορούν να αποφασίζουν για τα λιμενικά τέλη, τούτου δοθέντος όπως γίνεται στην Ισπανία, να λαμβάνουμε υπόψη πώς γίνεται αυτό, όπως στην Ισπανία, ε, στα πλαίσια των, που θέτουν οι εθνικές αρχές. Έτσι δεν θα απέχουμε και πολύ από το σύστημα που έχουμε και στους σιδηροδρόμους, όπου οι χειριστές των υποδομών έχουν μεγάλη ελευθερία, αλλά αυτή η ελευθερία κινείται εντός ενός εθνικού πλαισίου. Για το δυσκολότερο κεφάλαιο, το 2, ευπρόσδεκτος ο νέος προσανατολισμός του κυρίου Φλέκενστάιν. Εστιάζεται περισσότερο στη διοργάνωση των λιμένων, να θέσει ένα πλαίσιο στη διοργάνωση των λιμένων βασικά χορηγείται ελευθερία για την επιλογή ενός μοντέλου ελευθέρου ανταγωνισμού που θα ισχύει ο ελεύθερο ανταγωνισμό, αυτή είναι μία επιλογή. Η άλλη είναι να διοργανώνονται οι υπηρεσίε αυτέ βάσει αποκλειστικών δικαιωμάτων. Αλλά κάνοντα το αυτό, όπω και στου σιδηροδρόμου, υπάρχουν κάποιε υποχρεώσει που συνδέονται με τη χορήγηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Αυτό για λόγους ελέγχου και λογοδοσίας καταρχάς χορηγούνται μεγάλα ποσά από δημόσια χρήματα στους λιμένες, αλλά θέλουμε να αυξηθεί και η διαφάνεια για να μπορούμε να, να έχουμε χνηλασιμότητα σε επενδύσεις, κυρίως επενδύσεις που προέρχονται έξωθεν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεύτερη πτυχή που αφορά τη διαδικασία που θα πρέπει να περιγράφεται στον κανονισμό είναι η ασφάλεια δικαίου. Κάποιοι αναφερθήκατε σήμερα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι λιμένες για να τους αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια της νομολογίας, ακόμα και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Διαπιστώσαμε ότι προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα από αποφάσεις δικαστηρίου, διότι οι βάσεις των διαδικασιών, τα θεμέλια δεν καθορίζονται στην νομοθεσία. Για την πλοήγηση Υπάρχει διέξοδος μέσω των τροπολογιών που έχει υποβάλει μια ομάδα. Προβλέπει γενίκευση της πιστοποίησης του ε, πιστοποιητικού ε, του πιλότου για την πλοήγηση. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιείται σε αυξανόμενο ρυθμό στα λιμάνια. Οπότε θα εξισορροπήσουμε την ευαισθησία, τη μεγάλη υπάρχει την ασφάλεια από τη μια πλευρά, με τη δυνατότητα καμιά φορά όταν δικαιολογείται να υπάρχει μεγαλύτερη ε, λειτουργική ευελιξία που θα παρέχεται στους χρήστες. Το είπα και την προηγούμενη φορά, ευπρόσδεκτη είναι η προσθήκη για τις κοινωνικές διατάξεις. Σίγουρα το παρόν κύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά τις ιδέες που προευλήθησαν. Ίσως μία πτυχή είναι υποχρεωτική μετακίνηση των εργαζομένων, ίσως αυτό προχωρά πολύ μακριά υποχρεωτική απόσπαση, αλλά αυτέ οι ιδέες δεν επηρεάζουν το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εφόσον αυτές οι ιδέες συνδέονται σαφώ με λειτουργικέ βελτιώσεις εντό των λιμένων για την αξιολόγηση συνεπιών και αντικτύπου, να ξεκαθαρίσω ότι πιστεύουμε, αφού είδαμε στις διάφορες τροπολογίες, ότι η παρούσα διαδικασία για τη μελέτη αντικτύπου είναι αυτή που ισχύει, εκτό βέβαια από τι κοινωνικέ πτυχές. Αν θέλετε πραγματικά να προχωρήσουμε και να συμπεριλάβουμε συμπληρωματικέ πτυχές στα πλαίσια της αξιολογήσεως αντικτύπου, σίγουρα κάποια θέματα που αφορούν τι κοινωνικέ πτυχές που δεν συμπεριλήφθησαν στην αρχική πρόταση, θα έπρεπε να εξεταστούν αναλυτικά. Ο συσχετισμό με την οδηγία για τι εκχωρήσει, η, η πρόταση του κυρίου Φλέγκενστάιν δεν προσπαθεί να περάσει από την πίσω πόρτα την οδηγία για τις εκχωρήσεις, ούτε να την εξοδετερώσει. Δεν υπάρχει ούτε διπλασιασμός, ούτε αλληλεπικάλυψη εν συγκρίση με την οδηγία. Πρόκειται περί απλουστεύσεως. Στην αρχική πρόταση θεωρήσαμε ότι θα διοργανώσουμε τους διαγωνισμούς και τον ανταγωνισμό εντός του κειμένου που αφορά τις εκχωρήσεις και του σχετικού άρθρου και του πλαισίου και ο κ. Σάκενστάιν ακολουθεί έναν δρόμο που παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια αλλά και απλούστευση. Είναι απλούστερο να εφαρμοστεί από τους εμπλεκομένους φορείς. Άρα είναι λογικότατη η πρότασή του. Για την εξαίρεση κάποιων ε, λιμένων σας παρακαλώ να είστε προσεκτικοί. Μην επιβάλλετε αυθαίρετα διαφορές μεταξύ λιμένων Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων, πιστεύω. Και αυτή αυτό το πλαίσιο χρησιμοποίησαμε στην πρότασή μας. Όλο το διευρωπαϊκό δίκτυο. Όλο το δίκτυο, στο σφαιρικά. Αυτό συνεπάγεται ορθολογική ανάλυση του, της χωρητικότητας και το όγκο των εμπορευμένων αγαθών και τη γεωγραφική ισορροπία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος Τέλος, κλείνοντας, Πρόεδρε, απευθύνω έκκληση για, για μηχανισμό ενισχυμένης διαβούλευσης που προτείνει ο εισηγητής για να ε, μπορεί να υπάρχει και καλύτερη συμμετοχή και των εμπλεκομένων φορέων. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φλέκενστάιν. Εγώ από δική μου πλευρά, ε, θέλω να πω σε αυτά που μόλις τώρα είπε η Επιτροπή ότι το νόημα της όλης ιστορίας είναι εκεί όπου δίδονται οι συμβάσει παραχώρησης θα πρέπει να ισχύει η οδηγία περί συμβάσεων παραχώρησης. Όμως, όταν δεν είναι σύμβαση παραχώρησης, αλλά πρόκειται για εκμίσθωση, ε, τότε δεν εκεί στα περιπτώσεις δυνατόν από το παραθυράκι να φέρνουμε τη σύμβαση παραχώρησης ως προς τα τέλη λιμένων. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην τα βρούμε με τους Ισπανούς, αλλά ακόμα και αν δεν τα βρούμε εμείς θα τα βρει το Συμβούλιο. Άρα δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι και πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Τρίτον, Κιζένα, ε, μάλλον υπάρχει παρεξήγηση. Εγώ δεν είπα ότι δεν χρειαζόμαστε την αγορά. Αυτό που έχει σημασία και νομίζω όλοι συμφωνούμε από αυτού είναι ότι δεν μπορούμε ε, να εξαναγκάσουμε ε, αναγκαστικά να φέρουμε την πρότασή μας την αγορά και να αναγκάσουμε τα λιμάνια να οργανωθούν διαφορετικά. Τέταρτη παρατήρηση. Μπορεί κανείς να συμφωνεί, να διαφωνεί αν το θέμα της επικουρικότητας είναι σωστό ή όχι, αλλά κύριε Βαντάλεν ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει κανείς. Αυτό που είπατε εσείς. Δηλαδή ότι όσον αφορά τα εργασιακά θέματα ότι όλα μπαίνουν καλώς. Όχι, δεν μπαίνουν καλώς. Κάθε χρόνο μπαίνουν και χειρότερα. Και όσον αφορά την ευκαιριακή απασχόληση, παραδείγματος χάρη, ε, υπάρχουν κάποιες ε, περίεργες ε, ερωτήσεις της Κομισιόν ε, για να διασφαλιστούν κάποιες θέσεις απασχόλησης. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν μιλάμε για την διασφάλιση ανταγωνισμού στα λιμάνια, εκεί οι εργασιακές σχέσεις και οι προϋποθέσεις εργασίας παίζουν ρόλο. Είμαι σύμφωνος να το δούμε λιγάκι με τη διατύπωση, αλλά εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, ίσως με λιγάκι διαφορετική μορφή από ό,τι αναφέρεται τώρα στα χαρτιά, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημαίνουμε ότι ενδεχομένως θα προκύψει πρόβλημα ανταγωνισμού έτσι ώστε αυτοί που είναι αρμόδιοι να κληθούν να συζητήσουν μεταξύ τους. Τελευταία μου παρατήρηση. Αν δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τις ε, μαζικές εξαιρέσεις, block exemptions, δεν θα ψηφίσω ούτε εγώ για την πρότασή μου, θα την καταψηφίσω. Είναι εκβιασμός, ναι, εκβιασμός γνώση και έτσι να το εκλάβετε. Διότι κοιτάξτε, αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε να διαφωνήσουμε σε αυτή την Επιτροπή με κάτι το οποίο θα έρθει, θα έρθει από την πίσω πόρτα από το παρατηράκι και θα τα καταστρέψει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε δικαίωμα να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Ο συνάδελφος κ. Ρικέ μας παρέπεμψε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ ως κάτοικος του Αμβούργου συμφωνώ απόλυτα και μην ξεχνάτε και εμείς κάπου κάποια στιγμή την επόμενη δεκαετία ε, θα ζητήσουμε, θα θελήσουμε να είμαστε υποψήφιοι για Ολυμπιακού Αγώνε. Βέβαια, επειδή τρει φορέ αποτύχαμε, είμαι σίγουρο ότι θα αποτύχουμε και την τέταρτη. Δεν έχω καμία ελπίδα. Κατά τα άλλα, ε, άκουσα επένου, θέλω να πιστεύω ότι ήταν ειλικρινή, αγνή και ειλικρινή η επένη αυτή. Ευχαριστώ και εγώ τους και ηγητέ και επιτρέψτε να κάνω και εγώ μια παρατήρηση. Ξέρετε, ούτε και εμένα μου αρέσουν όλα. Πρόεδρος, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για εκβιασμό ή όχι, το δικαίωμα της ελεύθερης γνώμης και το δικαίωμα της ψήφου κατά συνείδηση, αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά αυτά τα στηρίζουμε όλοι ανεπιφύλακτα. Η ε, ψηφοφορία προβλέπεται για τις 10 ε, Νοεμβρίου, σε παρένθεση το είπα και πριν, υποαίρεση, to be confirmed. Θα το κρίνουν αυτό οι συντονιστές μας. Τώρα, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τους, ε, τους <laughs> προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Βάμντεκαν κατάφερε να έρθει εδώ ο εντελφή του, ο γαμπρός του, η νύφη του, είναι όλοι εδώ και κάθονται εκεί πίσω. Καλωσορίσατε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης που είναι η κατάσταση Μεσόγειο και η ολιστική προσέγγιση για τη Μεσόγειο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες. 104 τροπολογίες υπευλήθηκαν συνολικά και μια ψηφοφορία θα γίνει αύριο ήδη. Συνεργάστηκα με τους σκιώδες εισηγητές για να βρεθούν συμβιβαστικές τροπολογίες, συμβιβαστικής λύσης. Και ελπίζω ότι αυτές οι συμβιβαστικές λύσεις θα τύχουν τις υποστήριξεις αύριο. Για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα αυτή την γνωμοδότηση αρχές του καλοκαιριού. Και δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο ε, σημαντικό θέμα, πόσο πολύ θα είχε έρθει στα φώτα της δημοσιότητας αυτό το θέμα τους τελευταίους μήνες. Η το προσφυγικό, η προσφυγική κρίση είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα είναι προσωρινή, θα συνεχιστεί. Εξάλλου μεταναστευτικέ ροές προς την Ευρώπη ε, μόνο αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, υφίστανται ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν πρόκειται παρά να αυξηθούν εξαιτία τη κλιματική αλλαγή και πολλών άλλων λόγων. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε η γνωμοδότησή μας να εστιαστεί στο αποτελέσματα που έχει αυτή η προσφυγική κρίση και κυρίως οι ροές στη Μεσόγειο στο, στις μεταφορές. Φυσικά η γνωμοδότηση αυτή ήταν πολύ δύσκολο να συνταχθεί γιατί οι εξέλιξεις τρέχουν, η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε εβδομάδα. Και επίσης η κρίση πλέον δεν περιορίζεται μονάχα στην Μεσόγειο, την διαπιστώνουμε και στη Βόρεια Θάλασσα, την Ανατολή, στη Δύση, παντού. Και κατά την άποψή μου, οι επιπτώσεις που η προσφυγική κρίση έχει στις μεταφορές ε, στην Ευρώπη δεν περιορίζονται μόνο στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μεσόγειο, αλλά και σε άλλες περιοχές. Αναφερόμαστε επίσης στην ευθύνη των εμπορικών πλοίων, των κροζιερόπλοίων και για την συμμετοχή τους, στην ευθύνη που έχουν τα πλοία αυτά, να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης προσφύγων στη θάλασσα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο χρειάστηκε πολύ συχνά να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και δυστυχώς δεν υπήρχαν οι απαιτούμενοι πόροι διαθέσιμοι. Τα εμπορικά πλοία έχουν διασώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από την πλευρά τους οι πλειοκτήτες, οι πλοίαρχοι, τα πληρώματα είναι ξεκάθαροι ως προς τη θέση τους. Είναι ζήτημα ηθικής για αυτούς να σώζουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στο θάλασσα. Είναι επίσης ξεκάθαρο και από πλευρά διεθνούς ναυτικού δικαίου ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Επομένως δεν πρόκειται για μια υπηρεσία επιπληρωμή. Υφίσταται έτσι κι αλλιώς στον τομέα της ναυτιλίας ένα σύστημα ασφάλειας και επομένω δεν θα ήθελαν ένα ξεχωριστό σύστημα ε, αποζημίωσης οι εταιρείε υπάρχει ήδη ένα, ένα σύστημα που λειτουργεί. Αλλά ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων και το εύρος τους είναι τεράστιο και επίσης πολλές φορές ε, θέτει σε κίνδυνο τα πλοία που συμμετέχουν σε αυτές. Εμείς θα θέλαμε να αναδείξουμε μέσω στους γνωμοδότησής μας τα εξής ζητήματα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν οι αποτούμενοι πόροι για να διοργανώνονται αυτές οι επιχειρήσεις διέλευνας και διάσωσης στην Μεσόγειο. Το εμπορικό ναυτικό και άλλα πλοία μπορούν να συνεισφέρουν, αλλά η κύρια ευθύνη βαρύνει τα άλλους, τα κράτη. Είναι επίσης σημαντική η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης. Και επίσης θα ήταν σημαντικό να αξιοποιηθεί και η τεχνογνωσία που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Δυστυχώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εμπόριο ανθρώπων που είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση για τους διακινητές. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα πρέπει να είναι μια κοινή προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Πιστεύω ότι για να σταματήσει αυτό το εμπόριο ανθρώπων ε, που κάνουν κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων, ο τρόπος για να σταματήσει είναι να διευκολύνουμε και να ανοίξουμε νόμιμους οδούς μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους σχεδόν ε, συζητητές για τη συνεργασία, τους συναδέλφους που ε, συνεργάστηκαν και υπέβαλαν τροπολογίες. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση που θα είναι χρήσιμη για την ένα ψήφισμα άλλο που θα χρησιμεύσει στην Επιτροπή Λύπε που θα καταρτήσει την τελική γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Έκλεισε λοιπόν ο κατάλογος των αγοριτών. Ο κ. Λουίς Ντεγκράντες Πασκάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη στάση που τήρησε από την αρχή μέχρι τέλους. Ε, με χαρά άκουγε τις απόψεις των άλλων ε, για το θέμα αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και σαν πολιτικός μπορεί κανείς να πέσει εύκολα σε παγίδα και δεν έπεσε αυτή την παγίδα συνεργάστηκε στενά με τους σκιώδεις εισηγητές επί ενός θέματος που μας ενδιαφέρει όλους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η γνωμοδότηση μπορεί να συμβάλλει από πλευράς Επιτροπής Μεταφορών στην όλη προσπάθεια. Δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε αυτά που αναφέρονται στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή. Νομίζω ότι η στάση της ήταν άψογη. Και όπως είπα, ήταν ανοιχτή, άκουσε τις απόψεις όλων και έτσι καταφέραμε να πετύχουμε συμβιβασμούς που ικανοποιούσαν τους πάντες. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό δείχνει πόσο ευφυής ήταν η στάση της ε, εισηγήτριας, πόσο σοβαρή και πόσο αυστηρή. Υπάρχουν 15 ε, συμβαστικές τροπολογίες που αντικατοπίζουν αλληλεγγύη και την ευθύνη που ήταν θέματα τα οποία είχαν υπογραμμιστεί στην έκθεση της ΛΥΜΠΕ. Και είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σαν Ευρωπαίοι όταν αντιμετωπίζουμε δραματικές καταστάσεις. Ε, προφανώς εμείς περιοριστήκαμε στα θέματα που εμπίπτουν στη δική μας δικαιοδοσία. Συγγνώμη, αντί να προχωρήσουμε και να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Διότι έχουμε τις ε, τις πλειοκτήτες εταιρείες που έχουν καθήκον να παρέχουν βοήθεια σε ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και Ρωτήσαμε τι εταιρείε αν είχαν κάποιο πρόβλημα όσον αφορά αποζημιώσει, ασφάλεια κλπ. Και είπαν όχι, ότι το παρόν σύστημα ε, τις καλύπτει. Δεν θέλουμε να είμαστε καθολικότεροι του Πάπα, βασιλικότεροι του Βασιλέως. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα από εκεί που θέλουν εκείνοι να προχωρήσουμε. Η... Το να αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας που πέτυχε στους αρχικούς σκοπούς ε, και αν αναθέσουμε και άλλους στόχους χρειάζονται περαιτέρω πόροι. Εκεί θα ήταν το κατάλληλο βήμα για περαιτέρω διαπραγματεύσει. Αυτά. Αυτά έχω να πω. Καλή τύχη στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε, κύριε εισηγήτρια. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις επιτευχθεί σε συμβαστικέ λύσει και έτσι πιστεύω δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποστηρίξουμε τη γνωμοδότηση όταν θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κύρκος, παρακαλώ. Thank you, Chair. Αγαπητοί συνάδελφοι, η τρέχουσα προσφυγική κρίση έχει σοβαρέ επιπτώσει στο εμπορικό ναυτιλιακό τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κιλώνη, με την οποία συνεργαστήκαμε εξαιρετικά, όπω και του υπόλοιπου κοιόδη εισηγητέ, για τι συμβαστικέ τροπολογίε που καταλήξαμε, τι οποίε η Σοσιαλιστική Ομάδα θα στηρίξει στην αυριανή ψηφοφορία. Με αυτές τις τροπολογίες, τις συμβιβαστικές, μιλάμε για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις μεταφορές και τονίζουμε τη σημαντική συμβολή των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους σε επιχειρήσεις διάσωσης. Προτείνουμε λύσεις ώστε να απαλλαγούν τα εμπορικά σκάφη του δυσανάλογο βάρος που έχουν υπομειστεί, χωρίς να μελούμε την προτεραιότητα της ανθρωπιστικής πτυχής της κρίσης. Σκοπός μας είναι να μεταθέσουμε το βάρος ευθύνης στους πραγματικά υπεύθυνους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ίδια κράτη-μέλη. Τα εμπορικά πλοία δεν θα έπρεπε να αντικαθιστούν τι διεθνεί υποχρεώσει έρευνα και διάσωση των κρατών μελών στη θάλασσα και την ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάλληλη ευρωπαϊκή απάντηση. Επιπλέον, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο γιατί εμπορικά πλοία που βοηθούν εθελοντικά του μετανάστε μπορεί να υποστούν κυρώσει. Ζητάμε τα κράτη-μέλη να μην ποινικοποιούν αυτέ τι πράξει διάσωση και την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρηση οδηγία 2001 του 51. Τελειώνοντα, να πω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά αν δεν μειωθεί η ροή των ανθρώπων που περνάνε από τη θάλασσα για να φτάσουν στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να οδηγηθούμε στη μείωση του φορτίου που δέχονται οι εμπορικοί στόλοι. Γι' αυτό ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής και νότιας πλευράς της Μεσογείου και γι' αυτό ζητάμε να ενδυναμωθούν τα προγράμματα επανεγκατάστασης και να δημιουργηθούν νόμιμες ασφαλείς οδοί για τους πρόσφυγες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω ε, τους συγητές, ευησυγητές και οδησυγητές και χρησιμοποιώ με τις ευκαιρίες για να εκφράσω και εγώ εκ μέρους του ECR την υποστήριξή μου προς τις περισσότερες τροπολογίες. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού του τόσο σημαντικού θέματος και αυτό μάλιστα το κάναμε και μέσα στο πλαίσιο των αρμοντιτήτων μας τα εμπορικά σκάφη είναι δεσμευμένα να σώζουν ανθρώπους ε, στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό το προβλέπει το Διεθνές Θαλάσσιο Δίκαιο. Ε, οι τροπολογίες που έχω καταθέσει εγώ παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή την κατάσταση των εμπορικών σκαφών τα οποία δεν ε, αμείβονται οποτεδήποτε συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ενέργειες διάσωσης. Τουν έχουν απώλειες γιατί καθυστερούν και μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα στον τελικό του προορισμό με καθυστέρηση. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια αυτόματη, αυτόματος μηχανισμός αποζημίωσης, απλά θα πρέπει να έχει κανείς κατά νου ότι τα εμπορικά σκάφη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης υφίστανται ζημιές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να αποζημιώνονται. Σας λέω όχι αυτόματα αλλά με κάποιο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή τα εμπορικά σκάφη θα είναι πιο πρόθυμα να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ε, διάσωσης. Κατά τα άλλα ε, να σας πω ε, και ότι επιβιβάζουν περισσότερους επιβάτες από αυτούς που επιτρέπεται. Γιωσέ Νάσιο Φάρη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγητρία για την πάρα πολύ καλή δουλειά της, όπως επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι η προσέγγιση ε, είναι ιδιαίτερα περιεκτική και πράγματι μοιάζει να ενδιαφέρθηκαν να λάβουν υπόψη τους και τις ε, προτάσεις των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν 15 τροπολογίες. Εκτιμώ τη δουλειά όλων, κυρία της κυρίας ε, Κέλεν. Όσον αφορά το θέμα της διάσωσης στη θάλασσα και της ύπα της αρμοστίας ε, προσφύγων, νομίζω είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πρόκληση για όλους. Οι μετανάστες ε, είναι ανθρωπιστικό φαινόμενο το οποίο οφείλουμε ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας. Γι' αυτό εγώ σας λέω ότι θα υπερψηφίσουμε κάποιες ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι ότι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει και ότι θα έχουμε ε, καλή συνεργασία τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γκράντες και η κυρία Κίλεναν που μίλησαν για, την, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας στη Θάλασσα. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όπως ήδη αναφέρθηκε τα εμπορικά σκάφη δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις ευρωπαϊκές αρχές που είναι οι πρώτες που καλούνται να δραστηριοποιούνται οποτεδήποτε ξεσπάει η κρίση. Υπάρχει υποχρέωση ηθική νομική όλων μας να συμμετέχουμε με τους κατάλληλους και απαραίτητους οργανισμούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ο ελάχιστος δυνατός κίνδυνος για όλους όσοι εμπλέκονται. Ελάχιστος κίνδυνος και για τους διασώστες και για τους μετανάστες. Pass ICOD παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετικό έργο που έκανε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αν κοιτάξει κανείς και τις διάφορες τροπολογίε φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ξεφύγει. Και χαίρομαι που τελικά καταφέραμε να επικεντρωθούμε στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, δηλαδή τα ζητήματα μεταφορών. Βεβαίως τελικά κάποιοι δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να υποβάλουν τροπολογίες για ζητήματα Frontex κτλ. Θέματα τα οποία όμως θα έπρεπε να συζητηθούν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και ήδη θα ήταν δύσκολο να συμφωνήσει κανείς επί της ουσίας. Ας μην προσπαθήσουμε λοιπόν να εισάγουμε ε, διατυπώσεις σχετικές με τα θέματα αυτά στην γνωμοδότηση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την εισηγήτρια για τις διατυπώσεις τις οποίες κατάφερε να καταλήξει στις συμβιβαστικές τροπολογίες με τους σκιώδεις και τους λοιπούς συναδέλφους. Επομένως ας σταθούμε στα θέματα των μεταφορών, ας μην εμπλακούμε σε ζητήματα που είναι περισσότερο της αρμοδιότητας της Επιτροπής Θεμελιδών Ελευθεριών, όπως για παράδειγμα ο ρόλος της Frontex ή η συνεργασία με Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει, έχει δίκιο ο Το ζήτημα είναι ήδη πολύ περίπλοκο και ευαίσθητο και πράγματι υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με τα ζητήματα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, όμως είναι δύσκολο να μην αναφερθούμε σε ζητήματα πολιτικής μετανάστευσης και εμείς ως Επιτροπή ε, Μεταφορών γιατί συχνά ακούμε ε, τους ανθρώπους να, είναι, να μην μπορούν να ανεχθούν ε, τον αριθμό των πνιγμών των μεταναστών ε, στην ε, Μεσόγειο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αντιδράσεις για την αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην Ευρώπη σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο. και θα έλεγα ότι κατά την άποψή μας η πιο αποτελεσματική ε, πολιτική είναι εκείνη που εφαρμόζει η Αυστραλία από το 2003. Ε, Σε αντίθεση με επιχειρήσεις όπως ο τρίτον ο το Μαρενόστρου, κανείς πνιγμός στην Αυστραλία, πάνω από 300 πνιγμοί στην ε, Μεσόγειο. Επομένως βλέπουμε το σύστημα της Αυστραλίας λειτουργεί. Βεβαίως αναφέρεται η θεμελιώδης αρχή του ναυτικού δικαίου για την υποχρέωση της βοήθειας προς τους ναυαγούς. Αλλά σήμερα έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετική, μια διαφορετική κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε και εξαιρετικά μέτρα, τα οποία κατά μία έννοια είναι και προς το συμφέρον αυτών των ε, ε, φουκαράδων οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Πώς λοιπόν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να ζητήσουμε περισσότερο από τα κράτη-μέλη να κάνουν επικοινωνιακές εκστρατείες προκειμένου να πείσουν τους μετανάστες να μην προσπαθήσουν καν να έρθουν, τουλάχιστον να το γνωρίζουν ποιες ε, επιπτώσεις θα έχουν αν βρεθούν παράνομα στο έδαφος τους, για παράδειγμα το γεγονός ότι θα απελαθούν προς τρίτη χώρα, όπως το έχει κάνει η Αυστραλία, όπως το έχει κάνει επίσης η Ιαπωνία. Εάν χρειάζεται προσωρινή αναστολή της συμφωνίας του Σέγγεν, πιθανώς να χρειάζεται επαναφορά των εσωτερικών συνόρων, να καταπολεμήσουμε τους διακινητές, οι οποίοι είναι ε, ε, εγκληματίες και αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και δια της στρατιωτικής ποδού με στρατιωτική συμμαχία με τρίτες χώρες. Βεβαίως τα θέματα αυτά. Ε, το θέμα στο οποίο θα αναφερθώ τώρα δεν είναι τόσο θέμα της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά έχει μεγάλη σημασία η σχέση που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρίτες χώρες, ιδίως στη Μέση Ανατολή, για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Εμεί εδώ αναφερόμαστε περισσότερο στα ε, πλοία του εμπορικού ναυτικού τα οποία αναλαμβάνουν ένα σημαντικό οικονομικό ρίσκο και αυτούς θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι τροπολογίες τις οποίες υπέβαλα. Στόχος μου είναι να σταματήσουν αυτά τα ναυάγια στη θάλασσα και πιστεύω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι presidente. Sí, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, σημαντικές οι προσπάθειες που έκανε. Έλαβε υπόψη τις απόψεις μας. Κανονικά αυτή είναι η αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά και οι μεταφορές παίζουν ρόλο Άρα και εμείς μπορούμε να επιληφθούμε. Είναι επικίνδυνες οι μεταφορές που γίνονται αυτών των ανθρώπων με αυτά τα σκάφη που είναι ανασφαλή. Και τα μεταφέρονται με απαράδεκτο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά ακόμα και όταν μετακινούνται εντό τη Ευρώπη με τα ψυγεία κλπ. Άρα, εφόσον αφορά τις μεταφορές, μπορούμε και εμεί να γνωμοδοτήσουμε και να παρουσιάσουμε τροπολογίε. Γι' αυτό ευχαριστώ την συνάδελφο Κιλόνεν που στην ε, τροπολογία 14 δέχτηκε τους ασφαλείς διαδρόμους, μια ιδέα ε, που εξετάζεται και θα μπορούσε να παρουσιάσει με ακόμα πιο καινοτόμο τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα. Όσον αφορά τους ναυλωτές, εγώ συμφωνώ. Είναι θεμητό να βοηθάνε χωρίς να δέχονται αμοιβή. Δεν θέλουν να μπουν σε όλη την ε, διαδικασία ή μάλλον δεν θέλουν να δεχτούν ε, κάποια ενίσχυση, δεν θέλουν να μπουν στο κανονικό, στο τακτικό σύστημα ε, του ασύλου κλπ. Απλώ να παρέχουν τη βοήθεια όταν χρειάζεται. Κάποια πλοία αληφτικά και εμπορικά ε, πλοία είχαν αλλάξει θέση και είχαν ακόμα ε, αρνηθεί να δώσουν τη θέση τους στη Μεσόγειο. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Η τροπολογία μου υπαριθμών 5 που υπέβαλα ακολουθεί αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει ούτω ώστε να μην έχουν τα εμπορικά σκάφη την υποχρέωση να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές θα πρέπει να έχουν όμως την δέουσα υποστήριξη όταν παρέχουν βοήθεια και δεν θα πρέπει να αλλάζουν χωρίς να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες, ε, ρότα και πορεία γιατί μπορεί να σημειωθούν ατυχήματα. Πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην δημιουργηθούν αρνητικά φαινόμενα. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να χρονοτριβήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Ήταν πολύ καλή συνεργασία. Ήταν μια γνωμοδότηση η οποία ήταν καρπός κοινή προσπάθειας. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια που μου έδωσαν. Είμαι σίγουρη ότι θα προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και σας ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Η ψηφορία αύριο 9 η ώρα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα τη ε, διάταξη. διάταξης. Πρόκειται για το όλο πακέτο των ε, θεωρήσεων. Ο εισηγητή κ. Ε, Νοέ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής που μου ανέθεσαν το θέμα αυτό. Έμαθα πολλά πράγματα. Ολοκληρώσαμε ένα εξάμεινο εργασίας με τους συναδέλφους, επεξεργαζόμενοι το θέμα και ήταν άριστη η συνεργασία μας. Ε, οι συνεργάτες μου από τις διάφορες ομάδες με βοήθησαν πολύ και έπρεπε να είμαστε σε επαφή και με 15 οργανισμούς διμερός ή σε διάφορους σχηματισμούς γίνανε και διάφορες ε, επαφές, ε, ε, συνεδρίαση της Task Force για τον τουρισμό. Σε διάφορα σχήματα συζητήσαμε το ζήτημα για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο. Αυτό που θα ήθελα να πω τώρα και που το συζητήσαμε με εσά που είχατε παραστεί σε αυτές τις συζητήσεις της προετοιμασίας και τις προκαρα... προπαρασκευαστικές συζητήσεις να επαναλάβω κάποια στοιχεία εδώ. Μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι το παρόν σύστημα Schengen για τις θεωρήσεις, αυτό που ισχύει, μας οδήγησε σε απώλεια 6,6 εκατομμύρια τουρίστες από Κίνα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, από την Αφρική γενικά, από τη Βραζιλία, από τις χώρες αυτές, από τις αναδυόμενες οικονομικά χώρες. 6,6 εκατομμύρια πολίτες, ε, τουρίστες χάσαμε. Λόγω του αυστηρότατου και απειρχιωμένου καθεστώτος ε, του Σέγγεν. Ε, και είναι μέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή και τη μελέτη, την επόμενη πενταετία 130 δισεκατομμύρια ευρώ θα είχαν παραχθεί εάν κατά κάποιο τρόπο χαλαρώναμε το καθεστώς για τις θεωρήσεις ή ακολουθούσαμε πιο ορθολογική προσέγγιση για την χορήγηση των θεωρήσεων. Μιλάμε για πλούσιους ε, τουρίστες από τρίτες χώρες, οπότε η Επιτροπή μας ε, έχει ένα καθήκον από την σκοπιά των μεταφορών και τη σκοπιά του τουρισμού έχουμε θεμητό συμφέρον ε, να υποβάλουμε σχετικές προτάσεις και να γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας. Βέβαια, η Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών έχει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το πακέτο αυτό. Ελπίζω να τους πείσουμε όμως για την αναγκαιότητα που υπάρχει να επιφέρουμε αλλαγές, αυτές που προτείνουμε. Δύο είναι τα θέματα που τίθενται. Πρώτα απ' όλα είναι ο κόντεξ, ο κώδικας των θεωρήσεων. Έχουμε 43 τροπολογίες εδώ από τις πολιτικές ομάδες. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι κανένα κομμάτι του κειμένου δεν θα μπορούσε, είναι τέλειο και δεν χρειάζεται κάποια τροπολογία. Καταλήξαμε σε κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες και στη συνεδρίαση των σκιωδών την περασμένη εβδομάδα μπορώ να πω ότι καταφέραμε να πείσουμε τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Η έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ δημοσιεύθηκε έκτοτε, προτείνει σε κάποιες φάσεις ε, αλλαγές και η Επιτροπή Μεταφορών και αυτοί έχουν υποβάλει τροπολογίες και εμείς έχουμε υποβάλει, η ΝΕΣ έχει υποβάλει 7 τροπολογίες. Η πρώτη συμβιβαστική αφορά την αιτιολογική σκέψη 11 και 18 τις τροπολογίες που αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις. Εσείς που παρακολουθήσατε συζητήσεις το ξέρετε, αλλά ήθελα να τα επαναλάβω αυτά εδώ. Στις συμβιβαστικές λοιπόν αυξάνουμε από την περίοδο πριν την αίτηση από 12 μήνες την πήγαμε στους 18 μήνες Αρκεί μία θεώρηση στο χέρι για να μπορεί να ζητήσει κανείς τουριστική βίζα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ναυτικούς. Τα πληρώματα σκαφών, τα πληρώματα πλοίων. Μόνο οι ετούντες που έχουν μπει νόμιμα προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιλέξιμοι, έχουν δικαίωμα για τη συγκεκριμένη ε, βίζα. Μία άλλη αλλαγή, μία άλλη τροπολογία έχει στόχο να προσαρμόσει τη γενικά της εμπειρίας που έχουμε από τον υπόλοιπο κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κλάουντια Γκυλιάρα από το ΕΛΚ μας βοήθησε να το εξετάσουμε το θέμα. Αναφέρθηκε στη δυνατότητα και μιας πλατφόρμας ε, στο διαδίκτυο για την καταχώρηση όπου θα μπορούμε να προσφέρουμε τεχνική βοήθεια και αυτό το προτείνει μέσω τροπολογίας. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη για αυτή την προσέγγιση, για αυτό το θέμα. Η δεύτερη τροπολογία, εκ μέρους του ΕΛΚ, καλύπτει 15, την 36 και την 37. Αυτή η επιλογή του διαδικτύου της λύσεως online θα παρέχεται δωρεάν στους χρήστες και τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις δέουσες προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εν γέννη ζητώ την υποστήριξή σας για την αύξηση της διαρκείας των πολλαπλών ε, θεωρήσεων. Τροπολογίε 6, 7 και 8, σε αυτέ αναφέρομαι. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τριετία που θα πρέπει να αναφέρεται σαν περίοδο. Θα ήθελα να αυξηθεί σε πέντε αιτία. Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε τον αριθμό των επισκεπτών από πλευράς επιχειρηματιών θα ήταν κίνητρο για αύξηση των οικονομικών σχέσεων. Ελάχιστο τρία χρόνια, μέγιστο πέντε χρόνια αναφέρεται. Εγώ θα πρότεινα δέκα χρόνια σαν μέγιστο όριο για την πολλαπλή βίζα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια, διότι μόνο οι ετούντε οι οποίοι ήδη έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν επιλέξιμοι για αυτή την πολλαπλή θεώρηση, για το καθεστώς αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν αυστηρότερη προσέγγιση. Καταλαβαίνω το πώς σκέφτονται, αλλά δεν δέχομαι τις απόψεις τους αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε από το ECR υπευλήθησαν κάποιες τροπολογίες. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο στην ψηφοφορία, πώς θα τα πάνε οι τροπολογίες. Ευχαριστώ την κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα για τις πολύ χρήσιμες τροπολογίες που υπέβαλε. Αυτό ήταν το πρώτο πακέτο. Έχουμε 16 τροπολογίες για το άλλο πακέτο, για την άλλη δέσμη. νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σύντομοι ένα λεπτό το πολύ. Κοιτάξτε, Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, βέβαια εγώ δεν φταίω, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε γιατί αλλιώς δεν θα ξέρει κανείς τι να ψηφίσει. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο σκέλος του πακέτου που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα νέο είδος ε, θεωρήσεων. Κύριε Αγγιγιά, έχουμε μία κοινή τροπολογία και ελπίζω να γίνει αποδεκτή το θέμα αυτό το συζητήσαμε με ΜΚΟ και ε, επαγγελματικές ε, ενώσεις. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τη ΛΥΜΠΕ και ελπίζω να επικρατήσει αυτή η άποψη. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και τη συνεργασία. το θέμα δεν είναι για ένα λεπτό. Γενικά είπα να είμαστε σύντομοι. Θα έρθει επίτροπος και γι' αυτό θα είμαστε σύντομοι. Η κυρία, ο κύριος Ντέλη. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους ε, της συναδέλφου μου, ε, μου ζήτησε η συνάδελφός μου να σας... Ε, διαβάσω την ε, εισήγησή της γιατί είναι σκιώδης εισηγήτρια και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναντέλφους για τις προσπάθειές τους. Έχουμε δύο θαυμάσια έγγραφα. Ε, τα, από τη μία θέλουμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα το, της ε, εκδόσεως θεωρήσεων, από την άλλη θέλουμε να διευκολύνουμε και το θέμα της ε, έλευσης στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες, οι περισσότερες προβλέπουν την ε, απλούστευση διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων. Οι διευκολύνσεις αφορούν τα πληρώματα και άλλους που έρχονται νόμιμα στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι δυνατόν να εκδίδονται θεωρήσεις στα εξωτερικά σύνορα με ένα σύστημα online πριν έρθει κανεί στην Ευρώπη και έτσι θα μπορέσουν και οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν την έλευση των ετούντων. Επίσης να υπάρχει και μία νέα ιστοσελίδα εκεί να μπορούν ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση. Ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα και εμείς είμαστε απλά ένα βήμα πιο πίσω. Όσον αφορά τώρα τη νέα θεώρηση, τη θεώρηση touring visa όπως λέγεται, είναι η τουριστική βίζα, δίνεται δυνατότητα σε τουρίστες, σε συνταξιούχους, ε, ε, καλλιτέχνες και άλλους να ε, ζουν για ένα χρόνο στην περιοχή Σέγκεν, βέβαια να μην μένουν περισσότερο από 90 μέρες σε μία και μόνο χώρα. Και για την έκδοση αυτής της θεώρησης κρίνει το κράτος μέλος όπου τίθεται η πρώτη αίτηση απόκτησης θεώρησης. Είναι μια καινοτόμος διαδικασία γιατί έτσι ε, θα έρθουν περισσότεροι τουρίστες στην περιοχή Σέγκεν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να διαβάσω κι εγώ. Η Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια από τον συνάδελφο Νταν Ντόλτον, η οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί απόψε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του σκιώδης η θέση του, του ECR εκφράζω. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφοριακό το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να εξετάζονται πιο αναλυτικά οι οποιασδήποτε αιτήσει για θεώρηση. Έχουμε δύο προτάσεις όσον αφορά το σύστημα προεγγραφής και για τις θεωρήσεις στα εξωτερικά σύνορα, τις υποστηρίζουμε παραμένουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια ε, και τη πιθανότητα κατάχρησης αυτών του τουριστικών θεωρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο ε, της, ε, μετανα, των μεταναστευτικών ρόλων στην Ευρώπη. Θα θέλουμε ε, στο φάκελο τη αίτηση για μια τουριστική βίζα να αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενο ότι έχει τη δυνατότητα του οικονομικού πόρου να συντηρεί τον εαυτό του έτσι ώστε να αποφύγουμε την κατάχρηση αυτού του συστήματο. Επίση, όσον αφορά τα προξενία, μα ανησυχεί η συντόμευση των προθεσμιών που προβλέπεται, δεν είναι ρεαλιστική. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία μπορεί να κλείσουν το προξενείο τους και αυτό σημαίνει ότι η πίεση θα μεταφερθεί στο προξενείο μιας άλλου, ενός άλλου κράτους ε, μέλους. Συνολικά πάντως σας ευχαριστώ όλους για την ε, συμμετοχή και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία. Gracias, presidente. De manera breve para. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, θα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, το οποίο ήταν οδήγησε σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η στόχη και συμφωνούμε με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Συμφωνούμε ιδιαίτερα με τις τροπολογίες που αφορούν την online πλατφόρμα Συμφωνούμε επίση με τη Γενική Αρχή ότι ο κώδικα θεωρήσεων χρειάζεται επικαιροποίηση. Και επίσης να ε, προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχουν ταξιδιωτική ασφάλιση τα άτομα αυτά για οποιοδήποτε γεγονός ε, θέλει συμβεί. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά ε, στοιχεία από τη δικιά μας την πλευρά. Ναι. Eh, eh, Σα ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό έργο που έκανε και στις δύο προτάσεις που και οι δύο πιστεύω θα βελτιώσουν το σύστημα των θεωρήσεων έτσι ώστε να μην είναι ε, να μην δημιουργεί εμπόδια ούτε στους τουρίστες, ούτε στους φοιτητές, ε, ούτε σε άλλους επαγγελματίε, καλλιτέχνες και άλλοι που αναφέρθηκαν. Τροπολογία 22. Θα την αποσύρω, την τροπολογία 22, που αναφερόταν στο 18 μήνο, γιατί έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές ροές και αυτή η έκθεση είναι άκερη. Γιατί η Επιτροπή μας προστείνει μια νομοθεσία με την οποία κάποιοι υπήκοοι τρίτων ε, χωρών θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα στο χώρο Σέγγεν κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους το φιάσκο του Σέγγεν θα έπρεπε αντιθέτω να μα είχε κάνει να αναρωτηθούμε αν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική για την χώρο Σέγγεν. Εγώ πιστεύω ότι η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η επανασύσταση των ε, εσωτερικών συνόρων όσο συνεχίζονται αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα από την Αφρική και από την Ασία. Γιατί με αυτό το σύστημα το οποίο μας παρουσιάζεται σαν ένα σύστημα για να ε, ταξιδεύουν οι πλούσιοι ε, υπήκοοι των χωρών στην Ευρώπη, είναι στην πραγματικότητα ε, μια, πίσω, μια κερκόπορτα. Για άλλη μια φορά έχουν προδοθεί τα κράτη-μέλη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Προσπαθείτε όλο και περισσότερο να υποβαθμιστεί η λειτουργία των εσωτερικών συνόρων στον χώρο Σέγγεν προημοδοτείται οι επερεθνικές δομές και καταργούνται οι εθνικές δομές, ενώ τα κράτη-μέλη θα ήθελαν στην πραγματικότητα να πάνε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υιοθετώντα αντί να υιοθετήσει μάλλον αυτήν την έκθεση, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να καταψηφίσει όλες τις προτείνομενες αλλαγές στον κώδικα ε, για τις θεωρήσεις. Ε, δεν πρόκειται να σταματήσει πουθενά η Επιτροπή, όλο και θα κατατρώει τις αρμοδιότητες των, ε, κρατών μελών. Ο Τομπίες από την Κομισιόν, παρακαλώ να είστε σύντομος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τα άλλα μέλη ε, για την υποστήριξη και τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση για την ε, θεώρηση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, θα τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Θέλω μόνο να σας πω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, δεν θα περάσουν όλα απαραίτητα στο Συμβούλιο, άρα θα είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμβιβασμοί. Συμβιβασμοί πρώτα εδώ και μετά στη συζητήση στο Συμβούλιο. Για την ε, βίζα των τουριστών, εμείς ε, ε, είναι, θεωρούμε ότι είναι σημαντική. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και βάση περιπτώσει θα είναι σχεδόν αδύνατον ε, για ε, να ε, πάρουν για αυτό το θέμα της θεώρησης την Turing Visa Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και αύριο Κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας, οι πολιτικοί που συμμετέχουν ε, στις μεταφορές και στον τουρισμό προσβλέπουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εκεί αναφέρονται διάφορα επιχειρήματα και ένα πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Ορισμένοι από εμάς προέβαλαν το θέμα της μετανάστευσης, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν ας αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Εκεί που ζω εγώ, στην Ουγγαρία, στο νότιο κομμάτι της Ουγγαρίας, εκεί στα νότια ήταν το πιο φλέγον κομμάτι της ε, μετανάστευσης. Λίγο πιο κάτω στο ερχόντουσαν πάρα πολλοί μετανάστες, αλλά κανείς δεν ζήτησε θεώρηση, βίζα. Δύο διαφορετικά πράγματα λοιπόν. Το ένα έχει σχέση με τη θεώρηση, το άλλο με τη μετανάστευση και δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και θα ζητήσω αύριο την υποστήριξή σας. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχουμε την ψηφοφορία και τώρα συνεχίζουμε με τις συνεδρίες των συντονιστών και όσοι δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρία παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα.